Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συγνήσουμε τη συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω. Να σε ενημερώσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται στο ίντερνετ. Λοιπόν, το ένα, η ημερήσια διάταξη. Έγκριση της ημερήσιας διάταξη. Σε σχέση με την τελική εκδοχή της ημερήσιας διάταξης που κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου, Έχουμε δύο αλλαγές. Πρώτον, η ψηφοφορία για την έκθεση Μπάρμπαρα Σπινέλ για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης θα λάβει χώρα το απόγευμα στις 4.30. Θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρω ψηφοφοριών μετά την, έκθεση, ε, μετά την ψηφοφορία της έκθεσης Παύλου Ραντζέλ για το σχέδιο κανονισμού και των συνθήκων ε, όσον αφορά την ε, εκτέλεση των καθηκόντων του διαμεσολαβητή. Σας παρακαλώ να δεχθείτε αυτές τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Θα ψηφίσουμε λοιπόν δύο εκθέσεις το απόγευμα. Σπινέλη και Ράντζολα. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, δεν βλέπω να υπάρχουν. Θεωρώ ότι εγκρίθηκε η τροποποιημένη ημερήσια διάταξη. Δεύτερο θέμα. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Επειδή είμαστε πολύ λίγοι σήμερα το πρωί, θα κάνω όλε τι ε, ανακοινώσει μου το απόγευμα πριν συναντηθούμε με τον κύριο Φερχόφστατ. Να σας ενημερώσω για τα ξυστέματα. Πρώτα απ' όλα, ολοκληρώσαμε δύο τριμερείς διαλόγους ενώ είναι για την πρωτοβουλία των ε, πολιτών. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν. Ο τελευταίος τριμερής διάλογος έγινε στις 13 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Ήταν ο τέταρτος. Ήταν και ο κύριος Τίμερμαντς, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ο Υπουργός Μπόγκνερ Στράους ή Υπουργός Μπόγκνερ Στράους για δύο θέματα ε, είχαμε διαφωνίες για να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση. Η ελάχιστη ηλικία ε, από τις οποίες οι πολίτες μπορούν να στηρίξουν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και η άλλη ήταν ε, η ατομική συλλογή. Το σύστημα ατομικής συλλογής θέλαμε να αποσυνδεθεί η ηλικία στήριξης από την ελάχιστη ηλικία του δικαιώματος εκλέγην. Δεν μπορέσαμε να βρούμε, να βρούμε συμβαστική πρόταση. <clears throat> Δεν δέχονται τη δική μας πρόταση. Και τελικά λοιπόν συμφωνήσαμε σε ένα συμβιβασμό. Είπαμε ότι ο κανονισμός θα επιτρέπει και τις δύο δυνατότητες. Θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιλέξουν την ηλικία στήριξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών, την ελάχιστη ηλικία στήριξης και επίσης το κείμενο θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να θέσουν αυτό το όριο στα 16. Και είπαμε ότι στη διαδικασία αναθεώρησης θα υπάρξει συμπληρωματική αποτίμηση της διαδικασίας αυτής. Το άλλο θέμα, η ατομική ε, συλλογή, τα συστήματα ατομικής συλλογής, πολλά κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να το επιτρέψουν τώρα σε αυτή τη φάση. Δεν είναι δεθμενά να περάσουν στο συλλογικό σύστημα. Είπαμε ότι θα υπάρξει μια φάση σταδιακής ε, κατάργησης, τριετής ε, φάση σταδιακής κατάργησης της ατομικής συλλογής όταν θα αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός. Καλό αποτέλεσμα. Τώρα για την προστασία των δεδομένων για Σωστέ εκλογέ. Είχαμε το δεύτερο τριμερή διάλογο. <clears throat> Ολοκληρώθηκε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους συζητητές Βίλαντ και Μπρέσο. Πήγαν πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό για να μπορέσει να εφαρμοστεί κατά τις επικείμενες εκλογές Νομίζω ότι είναι λογική η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε για τα κυριότερα θέματα. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Σέφλιν και την κυρία Μπρέσο. Συγχαρητήρια γιατί τα καταφέραμε και δεν ήταν εύκολο. Όπως είπα για τον Brexit θα μιλήσω όταν θα είναι περισσότερο. Είχα μια συνεδρίαση της Κόζακ την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστι υπό την Ρουμανική Προεδρία και συζητήσαμε και την πολιτική συνοχή στα πλαίσια του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ήταν σημαντικό το θέμα να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι ανακοινώθηκε ότι η Ρουμανική Προεδρία θα συγκαλέσει μια διακοινοβουλευτική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης δεν θα είναι μια έκτακτη συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ, αλλά θα είναι μια διακοινοβουλευτική ε, συνδιάσκεψη που θα λάβει χώρα κάπου το είδα. Θα είναι πριν από τη συνάντηση στο Σύμπιου, αρχές Απριλίου. Δεν έχουμε ακόμη την ημερομηνία. Θα είναι δύο εκπρόσωποι ανακοινοβούλιο κοινοβούλιο άρα και δύο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το τελευταίο από πλευράς ανακοινώσεων είναι το σχέδιό μας για τη συμπερίληψη της διάστασης, της διάστασης φύλου, mainstreaming. Οι συντονιστές ενέκριναν αυτό το νέο πρόγραμμα εργασίας στις 21 Νοεμβρίου του 2018. Μετά το συζητήσαμε με την κυρία Μαγκίνες που είναι η αρμόδια για τα θέματα mainstreaming φύλου εκπροσωπεί την Επιτροπή μας στο δίκτυο του mainstreaming φύλου και λίγαν προσεχώς θα το αποστείλει στην Προέδρο της Επιτροπής Γυναικών που είναι αρμόδια για τη λειτουργία αυτού του δικτύου στο Κοινοβούλιο. Αυτές θα είναι Επίσης, το απόγευμα, όταν θα συζητήσουμε για τον Brexit, θα σας εξηγήσω και για την προετοιμασία των ευρωεκλογών στα πλαίσια του Brexit και την ενδεχόμενη παράταση ε, ισχύω του άρθρου 50 για την οποία δεν είμαστε ακόμη σίγουροι αλλά θα προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παρευρεθείτε λοιπόν και το απόγευμα Σημεία 3 και 4. Έγκριση πρακτικών. Για τις συνεδριάσεις. 11 Ιουνίου, 20 Ιουνίου, 11 Ιουλίου, 3 Σεπτεμβρίου, 24 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά περσινά. Είναι διαθέσιμα αυτά τα πρακτικά. Αν μέχρι το τέλος της συνεδρίας θα θεωρηθεί ότι ενεκρίθησαν. Και επίσης, δύο κοινέ συνεδριάσεις με την Τζούρι για την ε, ερμηνεία και εφαρμογή του, της Διοργανικής Συμφωνίας για καλύτερη νομοθέτηση και, αυτές, και τα πρακτικά αυτά είναι διαθέσιμα. Οι συνεδριάσεις έλαβαν χώρα στις 28 Μαρτίου και 25 Απριλίου πέρυσι. Είναι διαθέσιμα λοιπόν τα πρακτικά και όπως και προηγουμένως θα θεωρηθεί ότι ενεκρίθησαν αν δεν υποβληθούν ενστάσεις πριν το τέλος της συνεδρίασής μας αυτά και επειδή ο μόνο Χαουρέγγι είναι εδώ μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5 πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις αναλυτικές διατάξεις όσον αφορά την άσκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δικαιώματος Έρευνας που θα δικαστήσει την οδηγία του 1995. Πολύ σύντομα να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα αυτό το παρακολουθούμε από την αρχή της θητείας μας. Εξάλλου, το κληρονομήσαμε από την προηγούμενη θητεία. Στις 25 Απριλίου 18. Εγκρίναμε ένα κείμενο με το οποίο συμφώνησε και η Επιτροπή και η Σλοβακική Προεδρία ή μάλλον δεν συμφώνησαν τελικά, διαφώνησαν και τους απέστειλα μία επιστολή, ένα non-paper με μία νέα διατύπωση επί των προτάσεων ο Ραμόν σήμερα θα προτείνει περαιτέρω βήματα για να ξεκολλήσει το θέμα και δεν επιτύχαμε αυτά που θα θέλαμε μέχρι στιγμής λόγω της ε, αντίθετης τάσης του Συμβουλίου και δεν έχουμε και στήριξη της Επιτροπής. Οπότε ήταν μια επιπλέον δυσχέρεια. Νομίζω τότε τα υπόλοιπα μπορεί να τα πεις ε, Σύραμον για να μην τα λέω εγώ. Παρακαλώ, έχεις το λόγο για να ολοκληρώσει το ιστορικό και να μας μιλήσεις και για το μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι, δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες ε, πολλές σχετικά με την θλιβερή αυτή η ιστορία. Θέλω απλώς να εξηγήσω στους ε, συναδέλφους της ΑΦΚΟ ότι τέσσερα χρόνια μετά το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας σχετικά με τη δυνατότητα που θα είχε το Κοινοβούλιο να έχει ένα κανονισμό ώστε να διαχειρίζεται μία από τις πιο σημαντικές του αρμοδιότητες που είναι το δικαίωμα στην έρευνα. Και πρέπει να ομολογήσω εδώ την απογοήτευση και την αγανάκτησή μου και όλου του Κοινοβουλίου πιστεύω. Διότι δεν κατέστη δυνατόν να διαπραγματευτούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα. Κανονισμός ο οποίος μας υποχρεώνει να διαχειριστούμε αυτή την αρμοδιότητα, αυτό το δικαίωμα. Και αυτό είναι και το περιεχόμενο της έκθεσής μου. Που λέγει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να υψώσει τη φωνή του. Γιατί μετά από τόσο καιρό δεν κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε την εντολή της συνθήκης Λισαβόνας. Η κυρία Χούμπνερ θύμιζε όταν η υποσλοβακική προεδρία συμφωνήσαμε οι νομικές υπηρεσίες των τριών οργάνων να συνεργαστούν επί νέου κειμένου, επί του οποίου θα ήταν δυνατόν να διαπραγματευτούμε. Καθότι το προηγούμενο κείμενο υπό το φως της έκθεσης David Martin που είχε εγκριθεί από την προηγούμενη εντολή είχε πέσει πάνω στην διαφωνία, τη ρητή διαφωνία της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Και κάπως έτσι στήθηκε το ιστορικό αυτής της ε, απόκλησης, αυτής της διαφωνίας, ε, συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε σε ένα νέο κείμενο ανεπίσημο, ένα non-paper και αυτό κάναμε επί έξι μήνες. Οι νομικές υπηρεσίες οι τρεις συνεργάστηκαν για να συντάξουν ένα κείμενο επί τη βάση των συμφωνιών που υπήρχαν Και έτσι η Επιτροπή ΑΦΚΟ ανέλαβε να συντάξει ένα νέο non-paper για να το στείλει στα άλλα θεσμικά όργανα για να ξεκινήσει ένας νέος τριμερής διάλογος διαπραγμάτευση το οποίο απαιτεί το νομικό πλαίσιο. Χρειάζεται να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν ώστε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τον κανονισμό. Αλλά δεν έχει γίνει αυτή η διαπραγματεύση, αυτή η συζήτηση. Την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου συναντήθηκα με εκπροσώπους της Αυστριακής Προεδρίας για να καταλάβω κατά πόσον είχαμε ακόμα μια μικρή ελπίδα να συζητήσουμε σε αυτούς τους λίγους μήνες που έμεναν, απέμεναν. και οπωσδήποτε παρά την καλή τους διάθεση ήταν προφανές ότι δεν είχαν την εντολή να διαμορατευθούν. Διότι τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο δεν θέλει να αναλάβει αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν θα πάω σε τεχνικά ζητήματα τώρα, κατά πόσον εμπίπτουν ή όχι στη συνθήκη συγκεκριμένα σημεία. Αυτά είναι μια συζήτηση που δεν ακριβώς καταφέραμε να έχουμε, να κάνουμε τα τεχνικά. Και έχει φτάσει το σημείο που πρέπει γιατί να πούμε. Γιατί αλλιώ ε, θα πρέπει να σιωπήσουμε και να αφήσουμε το θέμα στο διηνικές. Αλλιώς πρέπει να αναλάβουμε μια πολιτική θέση και αυτό προσπαθώ να κάνω στην έκθεση που είναι αν θέλετε μια τελική μαρτυρία που θα μπορέσουμε να διαβιβάσουμε στους συναδέλφους επόμενης εντολής. Προσπαθώντας να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί σε αυτό το θέμα, σε αυτό το φάκελο. Υπάρχει επιχειρηματολογία βεβαίως από πλευράς των υπηρεσιών της Κομισιόν και του Συμβουλίου που λένε ότι τα δικά μας επιχειρήματα είναι υπερβολικά και ότι επικαλούμαστε αρμοδιότητα που δεν έχουμε κτλ. εγώ αυτό που σας προτείνω είναι να εγκρίνουμε σε αυτό το έργο εργασίας μία σειρά αποφάσεων που ε, διεκδικούν μία ελάχιστη πολιτική αξιοπρέπεια. Καταρχάς μία διαμαρτυρία ε, καταγγελία σε υψηλότερο επίπεδο. Και νομίζω ότι ε, η πρόεδρος της ΑΦΚΟ θα πρέπει να αποστείλει μια επιστολή στον πρόεδρο Ταγιάννη, εξηγώντα τι έχει συμβεί, ώστε να ζητήσει ε, επισήμως, μάλλον να υποβάλει την καταγγελία του επισημότατα σχετικά με το θέμα αυτό και την άρνηση Συμβουλίου και Κομισιόν να συζητήσουν. Επίσης είχαμε προετοιμάσει προφορικές ερωτήσεις, το είχαμε κάνει και στο παρελθόν, αλλά τώρα ίσως θα είχαμε την ευκαιρία αφού απαντήσει το Συμβουλίο και η Κομισιόν στις διάφορες ερωτήσεις που σας προτείνω, να μπορέσουμε να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα. Γιατί το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ε, θα ήταν αυτό που θα υποστήριζε αυτές τις προφορικές ερωτήσεις εντός των οποίων θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την πολιτική μας θέση στο θέμα αυτό. Επίσης αυτό που σας προτείνω είναι η νομική μας υπηρεσία να μελετήσει κατά πόσον πράγματι υπάρχουν οι δυνατότητες ε, υποβολής στο δικαστήριο για την έλλειψη συνεργασίας, πνεύματος συνεργασίας από πλευράς Συμβουλίου και Κομισιών. στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι ασθενείς οι νομικές βάσεις αλλά πρέπει με κάποιο επίσημο τρόπο η Επιτροπή αυτή να εκφράσει επίσημα και κατοχυρωμένα τη θέση μας και την διαμαρτυρία μας. Γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια ε, πολλοί συνάδελφοί μου έλεγαν πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Επαναλαμβάνω είναι ασθενεί οι νομικέ βάσεις μιας τέτοιας υποβολής προς το δικαστήριο, αλλά και αυτό περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που σας ε, παρουσιάζω. Επίσης, για το 226 που είναι το άρθρο τη συνθήκη Λισαβόνας, που διέπει την πρωτοβουλία που έχει το κοινοβούλιο για να, το κοινοβούλιο με για να υλοποιεί το δικαίωμά του αυτό. Οι ρητές τέτοιες διατάξεις που συμπεριλαμβάνει η συνθήκη είναι το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, της διαχείρισης των επιτροπών των εξεταστικών και η εκλογική νόμη. Αλλά εκ μέρους του Συμβουλίου και της Κομισιόν σχετικά με τη διαπραγμάτευση, η διάταξη αυτή εγκαθιστά, αν θέλετε, ένα ε, δικαίωμα αρνησικυρίας. Και ίσως θα ήταν και η οδός, νομικός μιλώντας, προς μια μεταρρύθμιση, μια επανεξέταση των συνθήκων, συγκεκριμένων δηλαδή τέτοιων διατάξεων. Επίσης εκφράζει, ε, εξηγεί την υποχρέωση που έχει το Συμβουλίο και η Κομισιόν να συζητούν το Κοινοβούλιο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ή στα πλαίσια διαφόρων ε, νομοθετημάτων και άλλων κειμένων που έχουμε για την ε, καλύτερη νομοθεσία κτλ. Όταν μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου ή της Κομισιόν οδηγούν σε μια κανονική νομοθετική διαδικασία στην οποία συμμετέχει κανονικά το Κοινοβούλιο με, την εκθε... με τις εκθέσεις του, με τους τριμερείς διαλόγους κτλ. Εδώ, αντιθέτως, σε αυ... στα πλαίσια αυτής διαδικασίας δεν εξηγείται ακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις, οι συγκεκριμένες και ρητές υποχρεώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν έναντι ή μάλλον στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο αυτής διαδικασίας. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε τι έγγραφα θα αφήσουμε στο κοινοβούλιο της ερχόμενης εντολής. Γιατί κατά τη διάρκεια της, ε, των ετών αυτών που πέρασαν, θεωρώ ότι πραγματικά βελτιώσαμε λίγο το κείμενο αυτό με τις επιτροπές εξεταστικές που είχαμε, έρευνας που είχαμε αυτά τα χρόνια Και νομίζω ότι η δραστηριότητα του Κοινοβουλίου τουλάχιστον με το τάξη 1, 2 και 3 με τα Panama Papers όπως και την, ε, ε, την Εξεταστική Επιτροπή για τις ε, εκπομπές των οχημάτων, των αυτοκινήτων ήταν θέματα, παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων έρευνας που είναι δικαίωμα του Κοινοβουλίου. αλλά το non-paper επί του οποίου αναφερόταν ο David Μάρτιν είναι ένα πληρέστερο κείμενο από αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου βελτίωσαν, συμπλήρωσαν αυτό το κείμενο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το κείμενο που πρέπει να αφήσουμε τώρα δεν θέλω να μιλήσω για κάτι σαν διαθήκη, αλλά εν πάση είναι μια παρακαταθήκη. Που η ΑΦΚΟ το 2019 θα αφήσει για τους μελλοντικού συναδέλφους. Διότι θα πρέπει να λάβει χώρα και θα είναι πιο ρεαλιστικό στην επόμενη εντολή να λάβει η χώρα αυτή επιτέλου η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Επίσης προτείνω μία σειρά πολιτικών εκδηλώσεων. Θα το προτείνω εγώ στις διάφορες πολιτικές ομάδες και αυτό λέει και το κείμενο. Εχθές συναντήθηκα με τον αρμόδιο επικοινωνία του Κοινοβουλίου διότι και εγώ δεν έχω επαρκή γνώσεις για να δω τι πρέπει να κάνουμε ώστε να επικοινωνήσουμε, να κοινοποιήσουμε αυτό το θέμα και προς την ε, κοινή γνώμη, προς το κοινό. Πώς θα μπορούσαμε να κινητοποιηθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να το θέσουμε στις πολιτικές ομάδες, στους Spitzenkandidaten, διότι εδώ μιλούμε ε, για θεμελιώδη δικαιώματα και αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. θα πρέπει να ενημερώσουμε και τα... να διαβιβάσουμε τα, τα στοιχεία αυτά στα μέσα ενημέρωσης. Ίσως προτάθηκε να διοργανώσουμε μια συνάντηση, ένα γεύμα με κάποιους εκπροσώπους σημαντικών μέσων ενημέρωσης, ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή και θα ολοκληρώσω Πρόεδρε λέγοντας ότι αυτό το κείμενο το επεξεργαστήκαμε με τον κύριο Σόλτ, την κυρία Παγάθα, ε, ε, όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων αυτό που σας ε, ε, υποβάλλω εδώ ε, συνοψίζει τη θέση όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω κάτι άλλο προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο σκιώδεις παρόντες για τους φιλελεύθερους. Είμαι είτε Ευχαριστώ. Όταν ο συνάδελφος Χάουρικη ξεκίνησε να εργάζεται. Γι' αυτό το θέμα που είχε κληρονομήσει από την προηγούμενη θητεία, είπα στους παρόντες συναδέλφους ότι ήταν ένα από τα πιο κατάλληλα άτομα για αυτή την τόσο δια... Ε, περίπλοκη διαπραγμάτευση. Γιατί το γνωρίζουμε εμείς, ε, η Ισπανία έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα στη σταδιοδρομία του. Ε, δεν θα επαναλάβω όσα είπε. Τον στηρίζουμε οι διάφορες πολιτικές ομάδες αυτή τη στιγμή εκφράζει την απογοήτευσή του, αλλά υπάρχει αναγκαιότητα να αναλάβουμε δράση σε πολιτικό επίπεδο. Όλα όσα ανέφερε τα στηρίζουμε. Όλα. Για παράδειγμα, το ότι θα πρέπει να μελετήσουμε τι δράση μπορούμε να αναλάβουμε, να γίνει μια μελέτη. Γιατί δεν υπάρχει πραγματικά ε, σωστή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της ε, παρούσης είχαμε μια σειρά από ενδείξεις που μας επιτρέπουν να κάνουμε ε, την καταγγελία, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε μια δουλειά επικοινωνία ε, γι' αυτό. Όντω, θα έχετε τη στήριξή μα. Δεν είναι δυνατόν. Που άλλα θεσμικά όργανα προβάλλουν τις δυνατότητές τους δράσεις, εμείς να περιορίζουμε τις δικές μας, αυτές που έχουμε. Όπως είπε και ο κύριος και ξέρουμε τι έγινε με τις διάφορες επιτροπές έρευνας. Αυτό πρέπει να υποθεί. Και θα πρέπει να προωθηθεί το θέμα στην επόμενη θητεία. Αλλά για να γίνει αυτό δεν πρέπει να σιωπήσουμε. Θα μας κοροϊδέψουν άλλα 5-6-7 χρόνια. Έχετε όλοι μας τη στήριξη κύριε Χάουρεγγι. Είστε μετρημένος άνθρωπος. Εφόσον φτάσατε σε αυτό το σημείο που λέτε ότι πρέπει να το κάνουμε, ορισμένοι που είμαστε λιγότερο μετρημένοι το αναμένουμε. Σόλτς για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες του, τις πολιτικές προσπάθειες διότι πολύ συχνά ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και συμφωνώ με τα όσα είπε ότι εμείς ως συνομοθέτες θα πρέπει να επιμείνουμε να έχουμε το δικαίωμα έρευνας. Θα συμφωνείτε όλοι πιθανότατα ότι το κοινοβούλιο αυτό πρέπει να ασχολείται με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλα τα γεγονότα, τα προβλήματα, τις ε, διαφωνίες ε, στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Είναι όλα αυτά τα πολιτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Και τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο έχουμε το δικαίωμα έρευνα για οποιασδήποτε εξελίξεις, προβλήματα, κακές εξελίξεις. Υποστηρίζω λοιπόν την προσέγγιση αυτή. Χρειάζεται να γίνει μια ε, ολοκληρωμένη, ε, ε, ολοκληρωμένος έλεγχος για τις εργασίες που έχουν γίνει για αυτό το αρχείο επί και βάσει της έκθεσης του εισηγητή και της ΑΦΚΟ. Δυστυχώ υπάρχουν καθυστερήσει, θα το επαναλάβω. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Πρέπει να συζητήσουμε πώ μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία ώστε να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Θα είναι το τελευταίο, το έσχατο βήμα αυτό, αλλά αυτό θα πρέπει να κληροδοτήσουμε εμείς ως Επιτροπή για το αρχείο αυτό. Υποστηρίζουμε επίσης ε, την Άλντε πλήρως όλες τις προτάσεις που έχουν υποβάλει. αλλά ίσως να αποτελεί και μια ευκαιρία να γίνει κάποιο πρωινό ή ενημέρωση τύπου ό,τι θέλουμε να το ονομάσουμε, ώστε να ε, προσελκύσουμε την προσοχή του κόσμου στις εργασίες της Επιτροπής ΑΦΚΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι ξέρετε ε, η διάσκεψη, η κομματική διάσκεψη του ΑΕΒΔ ε, στη Γερμανία, ενό κόμματο στη Γερμανία, στο EFD, συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του για τι ευρωεκλογέ το να διαλύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουν δηλαδή να πετάξουν στα σκουπίδια το νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να μην το λαμβάνουν υπόψη όλη τη διαδικασία ολοκλήρωση ε, και το Συμβούλιο. Είναι ένα πολιτικό πρόβλημα σημαντικό αυτό και θα πρέπει να πούμε σαφώς ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας, να επιμείνουμε ε, στα δικαιώματά μας ε, όπως θεσπίζονται στις συνθήκες και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές εξελίξεις. Να αναπτύξουμε και τα δικό μας δικαιώματα είναι μια ευκαιρία πολιτική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι μια ζωντανή διαδικασία και θέλω να είμαι σαφής εδώ ότι υποστηρίζουμε τον εισηγητή σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Τζο Ευχαριστώ πολύ το συνάδελφο Χαουρέγγι. Με πολύ ενθουσιασμό ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά θέματα που θέλουν πολλή δουλειά και σε αυτό το θέμα δεν έχουμε επιτύχει αυτά που θέλαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Τα κράτη-μέλη δεν μας παρέχουν αυτό το δικαίωμα, δεν μας το χορηγούν, πρέπει να το κατακτήσουμε. Και τώρα, εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση σε πολιτικό επίπεδο. Αναφέρθηκαν ορισμένα στοιχεία. Ένα πρωινό, για παράδειγμα, ποιους θα καλέσουμε, επιλεκτικά κάποιους δημοσιογράφους. Μπορούμε να κάνουμε απλώς μια συνέντευξη τύπου, μια κατάλληλη στιγμή όπου να προσκληθούν όλοι, όχι μόνο ορισμένοι που θα επιλέξουμε. τους οποίους μπορούμε βεβαίως ε, επιπλέον να ενημερώσουμε. Έχουμε επίσης δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και ένα ψήφισμα στην Ολομέλεια. Στην προηγική εκστρατεία τα κόμματα νομίζω θα μπορούσαν να προβάλλουν αυτό το θέμα. Υπάρχει κενό εδώ. Να γράψουμε ίσως και στους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων να αναφέρουν αυτό το θέμα. Κάτι που δεν υπάρχει πλέον στο κείμενο. Η νομική υπηρεσία και άποψη του δικαστηρίου. Θα το αφήσουμε αυτό για αργότερα ή να το αναφέρουμε και αυτό σαφώς, ότι θέλουμε. Θα μπορούσε να εκφραστεί το δικαστήριο επ' αυτού. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανένα άλλο το λόγο. Έχουμε δύο από το Συμβούλιο, εκπροσώπου Συμβουλίου, η κυρία Μόνα Στίγκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας δίνετε το λόγο. Μια σύντομη απλώς παρέμβαση για να σας πούμε ότι εμείς παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις ε, στο φάκελο αυτό αναγνωρίζουμε τη σημασία του για όλα τα θεσμικά όργανα. Έχουμε σημειώσει τη θέση που εκφράστηκε εδώ σήμερα. Θα ενημερώσουμε αντιστοίχως το Συμβούλιο και ως Προεδρία θα παρακολουθούμε διαρκώς το θέμα αυτό προκειμένου να εντοπιστεί μία λύση. Μία οδός προς τα εμπρός. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, με την ευκαιρία να σας πω ότι συναντήθηκα, είχα μια συνάντηση με, τους, ε, με την Προεδρία στο Στρασβούργο την ε, περισμένη εβδομάδα, γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι στις Προεδρίες. Είχαμε καλή συνεργασία σε καλό πνεύμα με τους εκπροσώπους των Προεδριών, αλλά υπάρχει αντίρρηση από συγκεκριμένα κρατημέλη από ό,τι φαίνεται. Θα ήθελα να ζητήσω από τον επικεφαλή της υπηρεσίας της Κομισιόν για τις σχέση με το Κοινοβούλιο, ο Σέρις Λεγκάλ, ή είναι κάποιος άλλος, ε, ζητώ συγγνώμη, ε, Μιχαλίνα Ζέμπα, λέει Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που δίνετε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη που ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Φόρτη, είναι στη Ρουμανία και ο προϊστάμενος επίσης λείπει. Ε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για όλη τη δουλειά ή στο φάκελο αυτό. Είμαστε έτοιμοι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε εφόσον λάβουμε μία πρόσκληση σε επίσημη διαπραγματεύση. Σε επίπεδο υπηρεσίας διαβιβάσαμε τις ανησυχίες που έχει η Κομισιόν με τον paper αυτό είχαμε συμμετάσχει σε όλες τις συναντήσεις και στην συνάντηση στην οποία αναφέρεται του Δεκεμβρίου ο εισηγητής μαζί με το Συμβούλιο και πάντοτε είπαμε ότι για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα επαρκές νομοθετικό μέσο το οποίο βεβαίως να σέβεται την αρμοδιότητα των τριών θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει, έχει θέσει κάποιες κόκκινε γραμμές στο θέμα αυτό. Εμείς το παρακολουθούμε στενά. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και πολιτικής φύσεως. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα ξαναδώσω τον, το λόγο στο Ραμόν, αλλά ο Χέλμουτ ήθελε κάτι προηγουμένως. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Άκουσα μόλις το Συμβούλιο και τις εξηγήσει ε, καθώς και την ερώτηση του Τζο Λάινεν και θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα θα πρέπει να λάβουμε μια σαφή απόφαση, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να πάμε στο δικαστήριο. Το έχουμε συζητήσει πολλάκις. Ξέρω ότι και από το ΕΛΚΟ ο κ. Βίλαντ, ο Σκιώδης, ε, είναι υπέρ αυτή της προσέγγιση. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, γιατί ακούμε ε, από κάθε Προεδρία ότι το λαμβάνει υπόψη, ότι είναι έτοιμη για διαπραγματεύσει, ότι υπάρχουν ε, κόκκινε γραμμέ κτλ, κτλ. Αλλά χρειαζόμαστε μία σαφή προσέγγιση για το ζήτημα αυτό και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε αυτό το δικαίωμα έρευνας ε, υπέρ του συμφέροντος των πολιτών. Πρέπει να πούμε σαφώς ποια θα είναι η προσέγγιση μας Ευχαριστούμε, Ραμόν. Ε, συγγνώμη. Μάικολ, επίση. Μάικ, παρακαλώ. Να πω απλώς ε, προς τον ε, Ραμόν, προς τον εισηγητή, ότι μεταξύ της ε, δυνατότητας του πρωινού για το τύπο ή τη συνέντευξη τύπου, καλύτερα η συνέντευξη τύπου και το συντομότερο δυνατόν, αλλά εν πάση τόσο είμαστε μαζί σας. Ραμόν, θα θέλαμε να σε ακούσουμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε και για, την προφορική, για τις προφορικές ερωτήσεις, αλλά θα έλεγα να το κάνουμε στην αρχή της ψηφοφορίας να είναι περισσότεροι συνάδελφοι παρόντες. Επίσης, ακούσατε τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Κομισιόν και θα θέλαμε να σχολιάσετε και την διαθεσιμότητά σας για νέα συνάντηση πρωτού ολοκληρωθεί η διαδικασία και δηλαδή να το έχουμε εγκρίνει και αυτό, όπως και την πρόταση που προέρχεται από όλους τους για τα, αυτά τα βήματα που παρουσιάσατε στο κείμενο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα εγκρίνουμε την κατεύθυνση αυτή, ίσως να έχουμε κάποιες ε, ε, προσαρμογές ας πούμε λεπτομέρειας. Η γενική κατεύθυνση θα είναι αυτή. Ναι, προεδρεός προς τα όσα αναφέρει η Προεδρία, το, το working document, ίσως να, έχει, να μην έχει επίσημα εγκριθεί στην ΑΦΚΟ, αλλά υποβάλλοντας ε, τις διάφορες εκδοχές του, θα έλεγα ότι η σημερινή του μορφή εκφράζει, εν πάση περιπτώσει, τη συμφωνία των ομάδων. Αποτυπώνει ναι θα ήταν απαραίτητη η έγκριση με ονομαστική ψηφοφορία για τις προφορικές ερωτήσεις που υποβάλλουμε για να είμαστε σίγουροι ότι οι πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν και αυτό το συγκεκριμένο ώστε να υποβληθούν αυτά τα προφορικά ερωτήματα την ερχόμενη εβδομάδα και για το, τα όσα είπε η Μάιτε και σε επίσημες και σε άτυπες συναντήσεις μπορούμε να έχουμε διάφορες επαφές με τον τύπο με τα μέσα ενημέρωσης έχουμε διάφορες δυνατότητες αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές το έγγραφο θέτει το θέμα της υποβολής της νομικές υπηρεσίες ε, της δυνατότητας αυτής διότι οι εκπρόσωποι των νομικών υπηρεσιών έχουν εκφράσει διάφορες αφιβολίες σχετικά με την νομική βάση που θα μπορούσε να έχει το Κοινοβούλιο για να στραφεί στο δικαστήριο για το θέμα αυτό. Σχετικά με την ε, συνεργασία που θα έπρεπε να έχει από τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Εν πάση περιπτώσει η παρουσίαση της πρότασης αυτής θα πρέπει να γίνει. Είναι κοινή θέση να γίνει αυτή η μελέτη. Και το θέμα θα πρέπει να το εξετάσει και η Επιτροπή Γιούρη που θα πρέπει να λάβει τις σχετικές αποφάσεις γιατί δεν εξαρτάται από μας ένα νομικό έγγραφο επί τη βάση του οποίου η Γιούρη θα αποφασίσει. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα από αυτό. Ως προς τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι Κομισιόν και Συμβουλίου δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Ε, ευχαριστούμε. Φυσικά η διαδικασία που θα οδηγήσει τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα την κάνει ο Πρόεδρος μετά από τη γνωμοδότηση της Γιούρη. Οπότε είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Από όσο κατάλαβα εγώ θα πρότεινα το εξή. Κατανοώ μετά τις δικές σας ε, εργασίες με τους Κιώδης ε, εφόσον δεν προτείνει κανείς τίποτα ε, για το τι να κάνουμε και η ΕΦΚΟ έχει εγκρίνει το δικό σας έγγραφο εργασίας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε. Ωστόσο δεν καταλαβαίνω τη δική σας ε, στάση όσον αφορά την πρόταση της Ρουμανικής Προεδρίας. Είστε ε, διατεθειμένος ε, να κάνετε κάποια συνάντηση. Μήπως συμφωνήσετε κάτι για το Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και χωρίς εμάς ώστε να διατηρηθεί αυτή η επαφή και για το μέλλον. Ίσως μια τέτοια συνάντηση να αποδειχθεί χρήσιμη. Μα πάντα είμαι διατεθειμένος να συναντηθώ αλλά η Ρουμανική Προεδρία δεν έχει διαπραγματευτική εντολή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όποτε θέλετε και σήμερα να συναντηθούμε με τη Ρουμανική Προεδρία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη της συνεδριά του Συμβουλίου δεν ε, επιτρέπουν στη Ρουμανική Προεδρία να, να συναντηθεί μαζί μα. Αυτό πρέπει να καταγγείλουμε. Δεν είναι θέμα Ρουμανική Προεδρία. Τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν στη Ρουμανική Προεδρία να διαπραγματευτεί μαζί μα. Εάν λάβει εντολή, ξεκινάμε και αύριο. Αλλά αν δεν έχει και παρόλα αυτά θέλει να με συναντήσει και πάλι να τους δω. Αλλά δεν θα προχωρήσουμε, απλώς θα κάνουμε ευχολόγια. Πρόεδρος, άρα παραμένετε ανοιχτή, ευχαριστώ, ανοιχτός, ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Είναι σημαντικό τμήμα του νομικού πλαισίου για την εργασία μας στο μέλλον αυτός ο κανονισμός. Ε, έχουμε όμως κάποια μηνύματα που μας λένε ότι μπορεί στην επόμενη θητεία το Κοινοβούλιο μπορεί να αξιοποιήσει πολύ συχνότερα τη δυνατότητα <coughs> επιτροπών έρευνας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να υπάρχει ένα πλαίσιο που να μας βοηθάει. Οπότε θα έχουμε απλώς την ψηφοφορία για τις ε, προφορικές ερωτήσεις. Ε, σε δύο λεπτά. Λοιπόν, κλείνω το θέμα αυτό. Ευχαριστώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή επίσης για τη συμμετοχή τους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Οι πολιτικές ομάδες θέλετε δύο λεπτά ή είστε έτοιμοι. Λοιπόν,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 ελέγξουμε τα μηχανήματα, άρχεται η ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, 7 συνάδελφοι δεν έχουν ελέγξει, δεν έχουν ψηφίσει. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα δοκιμαστικά. They were first discussed with the shadows. No one proposed any amendments, and then they were sent to everybody last Thursday. So they all, uh, mm-hmm. it's just to adopt. Okay, so we can, okay. we can close the vote. I understand. Πέρας ψηφοφορίας, από όσο κατάλαβα, όλες οι κάρτες λειτουργούν. Έχουμε απαρτή, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία επί των δύο ε, ερωτήσεων ε, με προφορική απάντηση προς συζήτηση με έτοιμα προφορικής απάντησης προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο με, ε, για το δικαίωμα έρευνα. Τι συζητήσει αυτέ συζητήσαμε, ερωτήσει αυτέ συζητήσαμε με του Σκιώδη, τι στείλαμε σε εσά την περασμένη Πέμπτη. Κανεί δεν σχολίασε. Οπότε μπορούμε να τι ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ένας είναι κατά. Ποιος ε, απόσχει. Ένας. Ε, οπότε εγκρίνονται και οι δύο ερωτήσεις. Και ο Ζωζέ μου λέει τώρα ότι το σχέδιο ψηφίσματος θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα. Είχα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Αλλά ίσω γνωρίζουμε ήδη το αποτέλεσμα. Ε, συγγνώμη, δεν μου υποβλήθηκε το αίτημα αυτό. Α, καλά, δεν είναι σοβαρό θέμα. Όπω ξέρετε έχουμε μόνο μία αποχή, οπότε όλα οι υπόλοιποι που, ήταν, που είναι παρόντες ήταν υπέρ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Γκέρκ Σέπφλιν που έχει την πρώτη ψηφοφορία, που έχει την πρώτη έκθεση που θα ψηφίσουμε, βρίσκεται καθοδόν να περιμένουμε λίγο. Μου επικυρώνει κάποιο ότι έρχεται πράγματι. Ή αλλιώ μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά. Υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο εδώ. Uh, Επειδή λοιπόν ο Γιώργη, ε, δεν, ο δεν είναι εδώ, προτείνω να κάνουμε την υλοποίηση των συνθήκων, των διατάξεων των συνθήκων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Συμφωνείτε? Ξεκινάμε με την έκθεση τη Μάιτα Παγκαζά Ορτουντούα με την εφαρμογή των διατάξεων των συνθήκων σχετικά με την ηθαγένεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το κείμενο, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Συμβαστική 4 υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 35. Ποιο είναι υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 41 μόνο οι and fight against corruption ως προσθήκη στη συμβατική 6 υπέρ κατά οι σοσιαλιστέ είναι κατά υπέρ μάλιστα εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά Α, μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 43 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Μία γκουε παραπάνω. Ωραία, όλοι ψήφισαν πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 48 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 48 Άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 10 προς 9 50 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 50 Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 51 υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται 53 υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται 57 υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται 55 υπέρ. Κατά αποχέ. Να ελέγξουμε την 55. Άρχεται ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται με 10 προς 9 συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ να ελέγξουμε την 63 υπέρ, αν έρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 9 προς 10 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 66 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 9 προς 10 67 υπέρ Ελκ υπέρ ναι κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ. Κατά. 69. Να ελέγξουμε την 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας δεν έχει ψηφίσει. Ξανά. Ξεκολουθεί να λείπει ένας, οπότε, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Κλείνουμε την ψηφοφορία εγκρίνεται 11 προς 9 70 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 70 έχω μπερδευτεί τώρα λέει η πρόεδρος είμαστε στην 70 ελέγχουμε την 70 κάποιοι δεν ψηφίζουν οπότε δεν, ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω ελπίζω να μην καθυστερούν τα μηχανήματα αλλά πρέπει να κλείσουμε. Εγκρίνεται 11 προς 10, 5, 16, όχι, καταπίπτει. Πάμε στην 71 υπέρ, κατά. Α, δεν, δεν ξέρω να ελέγξουμε την 71, γιατί αλλάζεται γνώμη κάθε λίγο και εκεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 10 προς 12. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 73 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 11 προς 11 74 υπέρ κατά να ελέγξουμε και την 74 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 11 προς 11 απορρίπτεται 75 υπέρ κατά νομίζω το ίδιο ας ελέγξουμε μήπως υπάρχει ένας που άλλαξε γνώμη 75 ελέγχουμε ηλεκτρονικά κάποιος δεν ψηφίζει επίτηδες νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω πέρας απορρίπτεται 3 προς 19 πως είναι δυνατόν δεν φαινόταν 76 υπέρ 76 υπέρ κατά οι σοσιαλιστές είναι κατά. Πώς να ξέρω, λέει ο πρόεδρος. Ας ελέγξουμε την 76. Εσείς ε, κάποιοι σηκώστε τα χέρια σας πολύ γρήγορα, κάποιοι άλλοι πολύ καθυστερημένα και τελικά δεν ξέρω τι γίνεται. Πέρας. 10 προς 12 απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά και πάλι σοσιαλιστές οπότε απορρίπτεται είστε κατά ωραία ωραία οπότε απορρίπτεται δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε 79 υπέρ κατά από όσο κατάλαβα το ΕΛΚ είναι κατά να ελέγξουμε την 79. Πέρας. 10 προς 12. Απορρίπτεται. 5-24. 5-24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος δεν ψήφισε, κλείνουμε την ψηφοφορία. 11 προς 10 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Φαίνεται να εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε την 82. Κατά συνείδηση. Πέρας. Εγκρίνεται 14 προς 7. 83 και 5 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται ε, η συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ. Κατά ας ελέγξουμε την 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 10 προς 12. Συμβεβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές. Και ε, το έλκυνε υπέρ. Εγκρίνεται. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Σοσιαλιστέ είναι υπέρ. Όχι. Συγγνώμη. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε σε τουλική σκέψη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 18 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 9 προς 13 συμβιβαστική ε, ο, συγγνώμη, τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομίζω. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Σοσιαλιστές νομίζω ήταν επίσης κατά. Ναι. Απορρίπτεται λοιπόν απλά. Ε, συγγνώμη που είμαστε. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στις ε, γνωμοδοτήσεις πέτη 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πέτη 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πέτη 12 υπέρ κατά Ε, οι σοσιαλιστές είναι κατά. Να ελέγξουμε νομίζω την 12. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά... So we are voting 12. 12 λοιπόν. Ξεκολουθούν δύο να λείπουν. Το κλείνουμε λοιπόν. 11 προς 10 ε, εγκρίνεται. Πάμε στη 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε B υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε ΙΤΑ υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται λίμπε J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε ομικρόν υπέρ οι σοσιαλιστές είναι κατά να ελέγξουμε την λίμπε όμικρον λοιπόν. Όχι, διότι δεν βλέπετε εσείς συναδελφοί, εγώ βλέπω. Εγώ, κοιτά, εγώ σας βλέπω και δεν είναι σαφές, ξέρετε. Όχι, βλέπω το ότι κάνετε ένα σήμα, κάποιοι έχετε ψηφίσει διαφορετικά, δεν ζητώ συγγνώμη. Ωραία, θα πάω πιο αργά. Λίμπε όμικρον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας, ψηφοφο... Πέρας ψηφοφορίας. 12 προς 10 εγκρίνεται. Λίμπε ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 11 υπέρ κατά α... Ζητώ συγγνώμη να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ζητά συγγνώμη πάλι. Δείχνετε διαφορετικά τα χέρια σας σε διαφορετικές στιγμές. Τι να κάνω, λέει η πρόεδρος. Γι' αυτό προτιμώ να ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 10 προς 12 απορρίπτεται. Λίμπε 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 14 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την Λίμπε 14 ηλεκτρονικά. Πέρας. 10 προς 12 απορρίπτεται. Λίμπε 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία πέρας 19 προς 3 υπέρ συγχαρητήρια εγκρίνεται Πάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Σέπφλιν. Πάμε στην έκθεση. Σέπφλιν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη μέσω των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Ονομαστική ψηφοφορία. Yeah, yeah, that's what I'm waiting for. Ναι, μα περιμένω. Περιμένω. Δεν εξαρτάται από μένα. Άρχεται η ψηφοφορία. So, one is not voting. Λοιπόν, λείπει μία ψήφος. Α, πέρας. 18 υπέρ, τρεις αποχές, συγχαρητήρια. Ωραία, ολοκληρώθηκε. You can't. So it's enhanced. It will be enhanced cooperation. Λοιπόν, ενισχυμένη συνεργασία. Αλλά λαμασού. Μα Α Αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε έτοιμοι. Ψηφίζουμε την έκθεση Λαμασούρ. 11 υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Δεκτή. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Α, όχι, εγκρίνεται. Αλλά θα ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 14. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 15 προς 7. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές. Α, να ελέγξουμε τη 16. Πέρας. Δεκτή. 14 ψηφί υπέρ. 8 κατά. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ α, καταπίπτει, καταπίπτει ναι 21 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ ελέγχουμε 25 άρχεται πέρας απορρίπτεται 8 ψήφι υπέρ 14 κατά 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ Κατά αποχή. Όχι. Ελέγχουμε. Την 27. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 29 με την προφορική τροπολόγησή της. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει, άρα την ψηφίζουμε τροποποιηθήσα την 29 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή λίμπε 2 μόνο το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή Λίμπε 3 υπέρ κατά ε, αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ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 Απορρίπτεται 10-11. 2 υπέρ κατά αποχέ. 3 υπέρ κατά αποχέ. δεκτή, 4 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχέ. δεκτή, 7 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Λίμπε D υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Γνωμοδοτήσεις. Λίμπε α. Α, όχι, είναι εκτός πεδίου εφαρμογής. Θα τι ψηφίσουμε εφόσον δεν είναι εντό του πεδίου εφαρμογή. Θέλετε να τι ψηφίσουμε. Όχι. Καλά. Δεν ψηφίζονται. Τελική ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. 18 υπέρ 2 κατά 2 αποχές. Ε, συγχαρητήρια. Α, ο κύριος Λαμασού θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επιβραδύνω τις εργασίες μου, αλλά ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστώ τους Κιώδης για το θετικό τους πνεύμα, όλους τους συνεργάτες από τη γραμματεία, τις ομάδες και τους προσωπικούς μου συνεργάτες. Και τονίζω ότι την τελευταία έκθεση που παρουσιάζω ενώπιον του Κοινοβουλίου, μετά από 24 χρόνια παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαίρομαι που γίνεται στην Επιτροπή Σταματικών Υποθέσεων, που κατά την άποψή μου ήταν πάντα σημαντικότερη από την Προεδρία σας, κυρία Πρόεδρε, και παρουσία των συναδέλφων, και για ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει σημαντικό μέλλον για το μέλλον της Ένωσης και ευχαριστώ πολύ. Yeah. Yeah, thank you, Alan. Ευχαριστούμε, αλλά φτάσατε την τελευταία στιγμή για να προλάβετε να υποβάλλετε αυτήν τη σημαντική έκθεση. Ελπίζουμε ακόμα να αλλάξετε γνώμη. Ξέρω, ξέρω, λέει η Πρόεδρος. Πάμε στην έκθεση της κυρίας Μπρέσο για την υλοποίηση των διατάξεων για την εξουσία του Κοινοβουλίου για άσκηση πολιτικού ελέγχου της Επιτροπής. Ε, ένα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ <clears throat> κατά. Όχι. Α, έχει καλυφθεί από τη συμβαστική. 35. Να ελέγξουμε για την 35 παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. 11-11 άρα απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 εγκρίνεται. 40 και 41. 40 και 41 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε για την 40 και 41. Δεν ήταν σαφές. Πέρας, απορρίπτονται. 12-10. 42 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ. Καταπίπτει 43. 44 λοιπόν υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ να ελέγξουμε τις 45 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 13-9, 46 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 47 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 50 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 50 παρακαλώ. Πέρας. 10-12 απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κόντι 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική της συζυγήτριας για την παράγραφο 13 για τη διαγραφή μάλλον του άρθρου 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 καταπίπτει 55, 56 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 57 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 58 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται, συμβαστική 4 <clears throat> υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 με προφορική δεν έχει κανείς αντίρρηση Ω τροποποιημένη λοιπόν να ελέγξουμε όμως. Να ελέγξουμε την 77 παρακαλώ. Περάσει εγκρίνεται 14-8. 78 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 83. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. 11, 11 άρα απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε και την 86 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορια Πέρα. Πέρας. 12-10 εγκρίνεται. Σημαντική 1 αιτιολογικές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται να ελέγξουμε ίσως την 4 παρακαλώ 10 12. 10-12 απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά, να ελέγξουμε και την 5. Πέρας, 12-10 εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά και την 6 να ελέγξουμε παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται 11-11, 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κοντ B β υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την κοντ β πέρασε εγκρίνεται 12, 9, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 17 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 11-11 πάλι. Απορρίπτεται. 18 υπέρ Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και τη 18. Την 18. Πέρασε. 10-12 απορρίπτεται. 19 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά οι σοσιαλιστές είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 25 παρακαλώ. Πέρας και απορριπτεται 10-12. 26 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Έχω την εντύπωση να, να ελέγξουμε τόσο πάνω. Σηκώνετε το χέρι σας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και δεν καταλαβαίνω αν είστε υπέρ κατά. Απορρίπτεται 9-12. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γνωμοδοτήσεις κοντ. Α, όχι, όχι, εκτός πεδίου. Εκτός πεδίου. Τώρα πάμε στην κον 34, όχι, καλύπτεται. Άρα, τελική ψήφος. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρασε. 18 με 4 αποχές συγχαρητήρια. Και πάμε στην τελευταία. Χρειάζομαι κάποιον από την γραμματεία. Λοιπόν, ε, ε, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου συμβαστική 1. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 6. Σωστά. Προφορική τροπολογία 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 6 τώρα. Καταπίπτει. 4. Υπέρ. Κατά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Μια στιγμή παρακαλώ. The five amendment, please, ah, to five, okay, Στην πέντε, παρακαλώ. Μπορείτε να παρουσιάσετε την προφορική τροπολογία. Ναι, θέλω να παρακαλέσω οι συνάδελφοι να δεχθούν μια προφορική τροπολογία που υποβάλαμε τελευταία στιγμή. Και ζητάω συγγνώμη. Σας μοιράσαμε ένα χαρτί όπου λέμε ότι πιστεύουμε ότι το σύστημα αυτό λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης και του χώρου της Ένωσης δεν θα πρέπει να μεταγραφεί ένα προς ένα στο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή είναι η τροπολογία που συζητήσαμε με την εισηγήτρια για να την εγκρίνουμε αν συμφωνείτε. Εκτός μικροφώνου κύριε Πρόεδρος. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβεστική 2 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη συμβιβαστική 2. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι δύσκολο. Ξαναζητά συγγνώμη, Πρόεδρος. Είναι δύσκολο. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 2. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 2. Πέρας ψηφοφορίας. 20 προς 2. Φαντάζεστε τι σύγχυση μου δημιουργεί αυτή η κατάσταση με τα χέρια που τα σηκώνεται σε διαφορετικές στιγμές και δεν έχω και τη μετάφραση και μερικές φορές είναι διαφορετικά. Τέλος πάντων, πάμε στη 10. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στην 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 22 ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας Ποιο είναι το αποτέλεσμα, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 11 προς 5. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 23, δεύτερο τμήμα. 23, δεύτερο τμήμα. 23, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κοιτάξτε σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Κατά 23 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 23 διότι είδα αποχή ε, δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει ακριβώς οπότε κάποιοι δεν ψηφίζουν επίκαιδες μάλιστα πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 26 υπέρ. Έπρεπε να το είχατε πει πριν, δεν ψηφίζετε, όχι μετά. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε τελειώσει δηλαδή με, την πρωινή, με το πρωινό τμήμα της συνεδρίασης και θα επανέλθουμε στις 3. Κλείνουμε λοιπόν. Δεν θέλει ο συνάδελφος. Α, εγκρίνεται 15 προς 4. Πέρας. Τέλος των ψηφοφοριών. Θα επανέλθουμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ.